hello everybody for our afternoon session. I hope till o'clock will be Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε πρέπει να έχουμε, ιδίω στα γυρατιά μας, πρέπει να έχουμε καλέ συνθήκε όσον αφορά τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Δεξιδιωτικών Παροχών Γι' αυτό και έχουμε την έκθεση του κυρίου Μπράιαν Χάγε, στον οποίο δίνω και τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και πρέπει να ξέρετε ότι κάθε μέρα φροντίζω για το μέλλον μας. Πρώτα απ' όλα, συζητήσαμε, όπως γνωρίζετε, για αυτά τα θέματα αρκετές φορές. Είχαμε και την δημόσια ακρόαση Είχαμε βέβαια και την ε, δημοσιοποίηση της δικιάς μου της έκθεσης. Σήμερα έχουμε διάφορες τροπολογίες να εξετάσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και τους σκιώδες εισηγητές που υπέβαλαν τροπολογίες αλλά και τους υπόλοιπους συναδέρφους. Έχουμε 737 τροπολογίες σήμερα στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πολλές θετικές ιδέες. Έτσι πιστεύω έχοντας εξετάσει τις οδηγίες και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε επικοδομητικούς συμβιβασμούς που θα βελτιώσουν την κατάσταση όσον αφορά την αγορά των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιδιωτικών παροχών. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι όλους τους συναδέλφους που συνεργάζονται μαζί μου για να καταλήξουμε σε μια πλήρη έκθεση με ευρεία βάση και τη συμφωνεί όλο μέσα σε επόμενες εβδομάδες. Το θέμα της σε πρόεδρε, ένα και δύο κυρίως. Δεν υπάρχουν πολλές τις τροπολογίες. Ξέρω ποια ήταν η θέση της Επιτροπής και του Συμβουλίου και εγώ παρακολούθησα και την ε, την κατάσταση όσον αφορά αυτό το θέμα και μπορώ σήμερα να πω ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία προκειμένου οι απαιτήσει ε, της ε, Solvency 2 να μην εφαρμοστούν στον IOPS. Ο κοινωνικός στόχος πάντως είναι ότι υπάρχει ένα στοιχείο πολύ βασικό σχέσης με τα ιδρύματα εξωτερικών παροχών κοινωνή συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε ως στοιχείο ότι υπάρχει. Και πολλές από τις τροπολογίες που προτείνονται στην έκθεσή μου έχουν να κάνουν με αυτό. Οι ευρωβουλευτές δηλαδή από όλε ε, τις πολιτικές ομάδες θέλουν να αναγνωρίζεται αυτή η σχέση στην τελική, στο τελικό κείμενο. Έχουμε επίσης πολλές ε, τροπολογίες για την διευθέτηση διασυνοριακών ιδρυμάτων εξωτερικών παροχών. Εδώ πρέπει να ξέρουμε πώς θα έρθουν τα εμπόδια στις ε, διασυνοριακές δραστηριότητες των ε, ιδρυμάτων αυτών. Πώς δηλαδή μπορούμε να βελτιώσουμε τις ε, διασυνοριακές δραστηριότητες ώστε να μην εμποδίζονται οι δραστηριότητε ενό ιδρύματο σε άλλη χώρα. Είναι θέμα εσωτερική αγορά. Θέλουμε μια εσωτερική αγορά που να λειτουργεί, που να υπάρχει οικονομία κλίμακο και για τις ταξιδοτικές παροχές και να έχουμε μια αντίστοιχη αγορά που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο και από αυτού προτείνω και εγώ διάφορες τροπολογίες. Τώρα για τις ε, απαιτήσει όσον αφορά τα στα σταξιδωτικών παροχών. Άλλοι θέλουν να αφαιρεθούν απαιτήσει, άλλοι όχι. Εδώ δηλαδή διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και το καταλάβαμε και από τις συζητήσεις και το βλέπω και στις τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Το δικό μου το καθήκον Πρόεδρε, είναι να πετύχω μια ισορροπία μεταξύ των δύο θέσεων. Ώστε οι διασυνοριακές δραστηριότητες να μην βλάπτουν τα ευρήματα σταξιδωτικών παροχών. Συνεργάζομαι τους κοιόδης συζητητές από αυτόν και πιστεύω ότι θα την πετύχουμε αυτήν την ισορροπία. Και για να συνδυάσουμε τις θέσεις των δύο πλευρών, αυτών που θέλουν τις απαιτήσει και από αυτών που δεν τις θέλουν. Τώρα, κατά τα άλλα, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε βασικές κατευθυντήριες γραμμές. Η δικιά μου έκθεση ήταν αρκετά μακριά από το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. εκείνη είχαν μια περιγραφική διατύπωση κυρίως. Ξέρω βέβαια ότι κάποιοι θέλουν να ενισχύσουν το στοιχείο που έχει να κάνει με την παροχή πληροφοριών. Οι περισσότερες πάντως τροπολογίες που μας έχουν φτάσει μέχρι τώρα θέλουν να υπάρχει ένα πακέτο αρχών στις κατευθύνσεις γραμμές. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πάντως μετά και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης που ακολουθεί την ίδια λογική αυτήν ακριβώς να ακολουθήσουμε με κάποια βέβαια ευελιξία ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερες τροπολογίες συναδέρφων προκειμένου να λειτουργούν καλά τα ευρήματα εξοδοτικών παροχών και να αποτελούν ένα μοντέλο προς το οποίο πρέπει να κατευθυνθούν όλες οι χώρες. Τώρα έχω μιλήσει με συναδέρφους για τροπολογίες που έχουν υποβάλει μονομένα συνάδελφοι που δεν είναι σκιώδεις. Να ξέρετε ότι τις εξετάζω, ότι είμαι ανοιχτό για να δω πώς μπορώ να τις συμπεριλάβω στο τελικό κείμενο. Θέλουμε να καταλήξουμε σε μια αξιόπιστη οδηγία, σε μια καλή πρόταση και πάνω σε αυτήν να έχουμε συζητήσεις με το Συμβούλιο. Είχαμε συναντήσεις με τους κοιόδες εισηγητές μέχρι τώρα και έχουμε καθορίσει ημερομηνίε για τον Νοέμβριο ώστε να βρεθούμε και να ενημερωθούμε καλύτερα. 1η Δεκεμβρίου, λέει το αρχικό χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής μας, η επόμενη ημερομηνία. Θα έχω τις ε, απόψεις των σχεδόν και των άλλων συναδέλφων, προκειμένου να με συμβουλέψουν πώς θέλουν να προχωρήσω σε αυτή την υπόθεση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ισκιώδης τώρα. Για τους σοσιαλιστές, κύριε Στάνκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή, τον Brian Hayes. Πράγματι, το βασικό είναι να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία και αυτό ακριβώ προσπαθούμε να κάνουμε. Πάντως, σημείο κίνηση για τους σοσιαλιστές είναι ότι τα περισσότερα ιδρύματα στρατιωτικών παροχών είναι κοινωνικά ιδρύματα με κοινωνική δράση και σε μια τριγωνική σχέση μεταξύ εργαζόμενων, εργοδοτών και κυβέρνησης. Και αυτή η αρχή πρέπει να απεικονίζεται στο κείμενο. Τώρα, συχνά ή κυρίω αποτελούν εθνική υπόθεση και η ευρωπαϊκή τους διάσταση έχει να κάνει κύρια με τις διασυνοριακές τους δραστηριότητες όταν υπάρχουν. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ορισμός για τις διασυνοριακές αυτές δραστηριότητες. Με την ουσία, δηλαδή να υπάρχει διαφορετική κατηγορία για τα διασυνοριακά ιδρύματα σταξιδωτικών παροχών που έχουν διαφορετικά προγράμματα. Πρέπει να υπάρχει αυτή η διάκριση λοιπόν ανάμεσα στα διασυνοριακά και τα μη διασυνοριακά ιδρύματα εξοδοτικών παροχών. Γιατί υπάρχουν ε, αυτά που δρούν εθνικά, που είναι τα περισσότερα, και μόνο λίγα δρούν διασυνοριακά. Άρα δεν πρέπει οι κανόνες που θα θεσπίσει η Ευρώπη για τις διασυνορικές αυτές περιπτώσεις να υποχρεώνουν σε συμμόρφωση όλα τα ευρήματα των εξωτερικών παροχών, ακόμα και εκείνα που δεν έχουν διασυνορικές δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση λειτουργίας τους όταν αυτή υπάρχει. Και στηρίζουμε τις κατεξουδότηση πράξεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, για τα διασυνοριακά, όπως σας είπα, συμφωνώ και καλό είναι να έχουμε ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα ιδρύματα αυτά, σε τρίτο Όταν υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση. Είναι μια άλλη τώρα ευρωπαϊκή διάσταση που δεν καλύπτεται και αυτή είναι το ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Όταν μετατοπίζεται το ίδρυμα από το ένα μέρος στο άλλο. Δεν έχουμε αντίρρηση αν μετακινούνται για τους σωστούς λόγους και όχι για τους λάθους λόγους, να αποφύγουν ανταγωνισμό για παράδειγμα. Ελπίζουμε η οδηγία αυτή να εξετάσει και το θέμα του ρυθμιστικού αρμπιτράζ. Όντω υπάρχουν πολλές τροπολογίες που αναφέρονται στους κανόνες. Όλο και περισσότεροι συμμετέχοντες ε, διαπιστώνουν την ε, προβληματική που υπάρχει για το γρήγορο κέρδος σε μικρό χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του ECR. Leslie Fox. Πρώτα, ευχαριστώ τον συναδελφό μας για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον φάκελο, καθώς και άλλους και οδησηγητάς, διότι νομίζω ότι γενικά καλά τα πάμε και υπάρχει αλληλοκατανόηση. Οι δικές μου τροπολογίες αναφέρονται στην ανάγκη της του σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, διότι δεν θέλω μια αναθεώρηση της, ε, της ε, οδηγίας IOP που να επιβαρύνει τις χώρες μέλη. Και ένας τομέας όπου κάτι τέτοιο μου φαίνεται ότι μπορεί να γίνει, το άρθρο 35 για την κατάθεση ε, για μια κατάθεση, για το depository δηλαδή. Όσοι θα θυμάστε, το Ενωμένο Βασίλειο έχει προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις στο δικό του συνταξιοδοτικό σύστημα και προβλέπει αυτοεγγραφή σε διάφορα συστήματα ώστε και τα χαμηλότερα εισοδήματα να ενταχθούν σε συνταξιοδοτικά συστήματα. Η συνολική καθολική χρήση depositories όμως θα καταστήσει δύσκολο το να δοθούν συντάξεις σε χαμηλού εισοδήματος μισθωτούς και δεν πρόκειται να αυξήσει την ασφάλειά τους. Επίσης, το άρθρο 5 να μην επιβαρύνει ιδιαίτερα τα συστήματα με λιγότερα από 100 μέλη. Υπάρχει κίνδυνος το συμβαστικό κείμενο, όπως είναι τώρα, να καταστήσει ε, μη οικονομικά βιώσιμα τέτοια μικρά συστήματα. Το άλλο είναι το Fully Funded Requirements, το άρθρο 15. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει δυσκολία να βρεθεί μια ισορροπία εδώ ανάμεσα στην ενίσχυση των διαμεροφιακών κινήσεων και στην αποφυγή του ρυθμιστικού αρμπιτράζ. Η συμβαστική τροπολογία προσπαθεί να αποφύγει την πλήρη εφαρμογή τη απέτηση για πλήρη χρηματοδότηση όταν συγχωνεύονται για παράδειγμα δύο συνταξιδοτικά συστήματα. Θα είναι όμω αδύνατο να φτιαχτεί ένα εξαντλητικό κατάλογο εξαιρουμένων δράσεων και κάποια συστήματα τελικώ θα μείνουν απ' έξω. Καλύτερα η απέτηση να ε, επιβάλλεται όταν δημιουργούνται νέα συνταξιδοτικά συστήματα και ιδίω για τα, για τα διαμεθοριακά. Ε, οι τροπολογίε μου για το άρθρο 77α και το 78 που έχουν καινοτόμο περιεχόμενο και ζητούν πρόσθετες δοκιμασίες επικορικότητας και αναλογικότητας μετά από την λήξη των διαπραγματεύσεων στους τριμερείς διαλόγους. Και αυτό προς το συμφέρον της βελτίωσης της νομοθεσίας. Θα γνωρίζουν οι άλλοι ευρωβουλευτέ ότι η κυβέρνηση του Ενωμένου Βασιλείου προχωρεί σε επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης μα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια από τι αλλαγέ που θέλουμε να δούμε να γίνονται είναι οι εξουσίες των Εθνικών Κοινοβουλίων να βάζουν φρένο σε προτάσεις που παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας. Για την ώρα έχουμε αυτά τα τέστη της κίτρινας και της κόκκινης κάρτας, αλλά αυτά δεν είναι άμεμπτα διότι εφαρμόζονται μόνο όταν εμφανιστεί η πρόταση της Κομισιόν και καμιά φορά ή πολύ συχνά εμφανίζεται, υποβάλλεται η πρόταση, πηγαίνει στο Συμβούλιο, έρχεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όταν περνά μέσα από τους τριμηρείς διαλόγους εμφανίζεται με πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε πολύ σοβαροί σε ό,τι αφορά τις δοκιμασίες επικουρικότητας και αναλογικότητας και άρα πρέπει να πιάνουμε τις προτάσεις όχι όταν βγαίνουν από την Κομισιόν, αλλά όταν βγαίνουν πλέον από τον τριμερή διάλογο. Και αυτό το στόχο έχουν οι τροπολογίες που σας προανέφερα. Μην ευνηδιαστείτε εάν κάτι παρόμοιο έλθει και από την διαπραγματευτική ομάδα του Ενωμένου Βασιλείου. Θα ήθελα να ολοκληρώσω, ευχαριστώ τον Μπράιαν, ε, επίσης, ε, να ολοκληρώσω μάλλον, με ευχαριστήσει πάλι προς τον Μπράιαν για τον τρόπο που χειρίζεται το ε, θέμα τώρα. Σας ευχαριστώ, Άσλι, Φιλελεύθερη. Η κυρία Γκουλάρ δεν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ενωτική αριστερά. Ρουμπέν Κρέσπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, Όπω έχουμε πει από την αρχή, για μια αγορά πολύ εσωτερικευμένη και με έντονο εργατικό δυναμικό θέλουμε να διασφαλίσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα, να υπάρχει κινητικότητα και να καλύπτεται από τα κοινωνικά αυτά δικαιώματα για τους εργαζόμενους που μετακινούνται. Να υπάρχει διαφάνεια και να διευκολύνεται η ενημέρωση των εργαζόμενων ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να μπορούν να τα υποστηρίξουν. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιηθεί αυτό λοιπόν ως μια ευκαιρία για κερδοσκοπικές και επικίνδυνες δράσεις. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνούμε με τους πράσινους για το ότι πρέπει να γίνουν μελέτες για τους κινδύνους επί του περιβάλλοντος των επενδύσεων αυτών. Γιατί οι αποταμιεύσεις μας δεν πρέπει να χρησιμεύσουν για να επιδεινώσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση του περιβάλλοντος. Τα συνταξιδιωτικά ιδρύματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα κοινά αγαθά, το δημόσιο χρήμα για στραβούς σκοπούς οι επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση των λιμένων ή άλλων ενεργειακών υποδομών, υποδομών μεταφορών. Τα στρατιωτικά συστήματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται πλήρως. Για μας αυτό είναι βασικότατο, διότι πιστεύουμε ότι είναι κοινή λογική. Αλλιώς παίζουμε με το μέλλον των εργαζόμενων και με τα δικαιώματα των ε, δικαιούχων συντάξεων. Δεν πρέπει να γίνεται κερδοσκοπία. Δεν πρέπει να εξαρτάται από την κερδοσκοπία ε, το, μέλος, το μέλλον των ε, συνταξιούχων. Συμφωνούμε λοιπόν με την πρόταση των πρασίνων. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ ανησυχητικό που δεν δέχεται τις εγγύησεις εφαιρεγγιότητας για αυτό το Ταμείο Συγητής. Εμείς δεν θέλουμε να μειωθούν οι απαιτήσει σε κάτι τόσο ζωτική σημασία όπω είναι οι συντάξει. Δεν στηρίζουμε λοιπόν την οδηγία για την φερεγκιότητα, αλλά το να επιτρέψουμε να υπάρχουν λιγότερες απαιτήσει φερεγκιότητας για αυτά τα ευρήματα θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κερδοσκοπία όπου οι ενδιάμεσοι θα υποφεληθούν για να κερδίσουν περισσότερο από τι επενδύσει. Κυρίε και κύριοι, οι συντάξει είναι βασικό δικαίωμα. Δεν είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να παίζουμε, να κερδοσκοπούμε. Δεν μπορούμε να παίζουμε στο καζίνο με το δικαίωμα στη σύνταξη του κόσμου. Το έχουμε κάνει πάρα πολύ καιρό και τώρα ακριβώς αυτό πληρώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Φέρβερ, σας ευχαριστώ. Ο σκιώδης ηγητής των Πρασίνων δεν είναι παρόν, αλλά λαμβάνει το λόγο ο αρχηγός τους. Φίλιπ Λάμπερτ, σας ευχαριστώ Μάρκους. Χθε ήμουν Μισελ Λεϊμόν, σήμερα ε, το πρωί ήμουν άλλο συνέδελφο, Σβεν Γκίγκολτ, σήμερα πάλι το απόγευμα. Τέλο πάντων, παίζω πολλού ρόλου. Ποιο είναι το κόνσεπτ, η βασική ιδέα, διότι πρόεδρο ομάδο για εμά του πράσινου είναι ο υπηρέτη των υπολείπων. Να τον αντικαταστήσετε αμέσω λέει ο πρόεδρος. Μάλιστα, λοιπόν, εγώ λοιπόν κάνω όλη τη δουλειά εδώ, εδώ το management κάνει τη δουλειά και αυτοί βρίσκονται επί τόπου, στο πεδίο, για να βρουν καινούριου ψηφοφόρου, α το πω έτσι. Για την AOP. Πρώτα για την διαφάνεια. Αυτό που θέλουμε είναι οι δικαιούχοι να γνωρίζουν πού πάνε, τι γίνεται με τα μελλοντικά τους χρήματα. Ποιες εγγυήσεις έχουν δηλαδή από τις ε, συντάξεις του δεύτερου πυλώνα να αυξηθεί η διαφάνεια στην επενδυτική δραστηριότητα των ταμείων, ώστε να γνωρίζουν οι δικαιούχοι πού επενδύονται τα χρήματα των συνταξιωτικών ταμείων. Άλλο σημαντικό για μας είναι όχι μόνο η διαφάνεια σχετικά με τις μελλοντικές απολαβές, αλλά να γνωρίζουν και τον ενδεχόμενο κίνδυνο που επιφέρουν οι επενδύσεις, δηλαδή ποιο είναι το σενάριο, το χειρότερο ενδεχόμενο σενάριο να είναι προετοιμασμένοι οι άνθρωποι και να έχουν κάποια ορατότητα σχετικά με το τι γίνεται και ποιους κινδύνους, σε ποιους κινδύνους εκτίθενται. Θα θέλαμε επίσης να συμφωνήσουμε στο ότι κάποιο streamlining ε, της προτάσεως της Κομισιόν είναι αναγκαίο για τα AOP όσο αυτοί οι εφόσον δηλαδή οι στόχοι της διαφάνειας δεν ε, υπονομεύονται. Βεβαίως και πρέπει να είναι πλήρω χρηματοδοτημένα, fully funded, το πιστεύουμε εμείς αυτό, και δεν βλέπω για κανένα λόγο γιατί όχι. Μιλούμε για σόφρονα διαχείριση, έτσι δεν είναι. Και επίσης δηλώνουμε ότι μας εκπλήσει το γεγονός ότι πολλά από τα ταμεία αυτά υποθέτουν ότι θα έχουν κέρδη από τις επενδύσεις τους όχι μόνο μη ρεαλιστικά αλλά και πολύ περισσότερα και από αυτά που αναμένουν πολλές ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Οι Ολλανδικές τράπεζες έχουν βγάλει μια έκθεση που λένε ότι είναι απολύτως μη ρεαλιστικά. 4% αναμένουν μακροπρόθεσμα οι τράπεζε του συμβουλεύουν να μην αναμένουν παραπάνω από 3,3% και ήδη και αυτό εμένα μου φαίνεται κάπως υπερβολικό. Θέλουμε λοιπόν συντηρητική διαχείριση και με την έννοια αυτή κύριε Φέρμπερ συμπαρατασσόμεθα μαζί με εσάς τους συντηρητικούς, είμαστε συντηρητικοί και εμείς για το ε, χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και είμαστε συντηρητικοί και τον πλανήτη, συντήρηση θέλουμε να διατηρηθεί δηλαδή. Γι' αυτό είμαστε πράσινοι. Θέλουμε λοιπόν αυτές οι προειδοποιήσεις να ληφθούν υπόψη άλλου είδους προειδοποίηση που είδαμε από ένα Καναδό, ο οποίος είναι επικεφαλής της Τράπεζας της Αγγλίας, μακάρι για τον οποίο έχουμε και πολύ μεγάλο σεβασμό, είναι για τα περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία του ενεργητικού, που ε, προκύπτουν από ορισμένε επενδύσεις που αναφέρονται στην ε, φούσκα του διοξιδίου του άνθρακος. Carbon bubble, λέει ο ε, κ. Λάμπερτ. Ε, που έχουν ε, επενδύσει πάρα πολύ ορισμένοι. Θα πρέπει λοιπόν μακάρι και άλλοι να εισακουστούν αξιοσέβαστη προσωπικότητα που ηγείται ενός αξιοσέβαστου οργανισμού και που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Άρα πρέπει να ισχύσει και εκεί σοφροσύνη και να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία αυτά και στους υπολογισμούς των κινδύνων που αναλαμβάνουν τα συνταξιδοτικά ταμεία. Τώρα, ακόμα ωστόσο και ένα όργανο, ένας οργανισμός, ο οποίος ε, γίνεται αντικείμενο καλής διαχείρισης, μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες εφόσον πέσει σε μια κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο να επιτρέψει την ανάκτηση ή την ανάκαμψη και όχι το ξεπούλημα. Να μπορεί δηλαδή να χειριστεί τα πράγματα σωστά εφόσον πέσει σε ταραγμένα ύδατα. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις που κάνατε και για τα όλα τα υπόλοιπα σχετικά τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Τώρα, η ομάδα EFDD, ο κύριος Βάλι. Ευχαριστώ Πρόεδρο και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές, διότι διάβασα τις τροπολογίες του και οφείλω να πω ότι σίγουρα το κείμενο θα είναι καλύτερο από αυτό που πρότεινε αρχικά η Κομισιόν. Καλύτερη διακυβέρνηση, καλύτερη διαφάνεια, διαχείριση του κινδύνου. Συμφωνώ. Καταρχήν όμως θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ πριν αφήσουμε να σειρεύσουν οι ε, ε, συμβολές, αυτά τα ταμεία, ε, στον ε, τομέα το χρηματιστηριακό, γιατί εκεί υπάρχουν προϊόντα πολύ επικίνδυνα. Θα πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι στην πράξη την οικονομία δεν την έχουμε εξωτερώσει, ο συστημικός κίνδυνος είναι σημαντικός, σημαντικές διατάξεις όπως η BSR ή η ρύθμιση της σκιώδους τραπεζικής έχουν περάσει σε δεύτερο πλάνο σε αυτή τη διάταξη και μπορεί να πληρώσουμε τις συνέπειες εάν υπάρξει κρίση που μπορεί να προκύψει και λόγω εξωτερικού ε, παράγοντα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη, το ευρώ θα πρέπει να είναι έτοιμο. Ίσως τώρα να μην το σκεφτόμαστε και να προχωράμε με σκημένο το κεφάλι προτείνοντας διατάξεις που τελικά οδηγούν στην ίδια κατεύθυνση όπως την προηγούμενη θητεία. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ. Έχουμε υποβάλει προτάσεις για τα δεξιτικά ταμεία βέβαια που θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται πλήρω, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι πριν από μένα και θα πρέπει να επενδύουν με στόχο μακροπρόθεσμο και όχι βράχη πρόθεσμο. Δηλαδή όσο γίνεται λιγότερη κερδοσκοπία και να λαμβάνεται υπόψη και ο κοινωνικός αντίκτυπος αυτών των επενδύσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί διαφορετικά η ρευστότητα πάει σε επενδύσεις με κερδοσκοπικό στόχο και δεν ε, λαμβάνει κανείς υπόψη το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πλήρης απαγόρευση λοιπόν να χρησιμοποιούνται μέτρα τα οποία δεν είναι ρυθμισμένα, δηλαδή που ε, ε, είναι αδιαφανή και πολύ κειμενόμενα. Να φροντίσουμε λοιπόν ώστε αυτό το σχήμα να είναι απόλυτα διαφανές ε, για όσον αφορά τους επενδυτές και ε, δημόσιο ε, το ότι κάνουν αυτά τα ταμεία έτσι ώστε να γνωρίζουμε τους κινδύνους, να είναι εγγεγραμμένα τα κριτήρια απόδοσης που χρησιμοποιούν, τα κόστη, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, αλλά και όλες, όπως είπα, οι πληροφορίες αυτές να είναι δημόσιες και διαφανείς. Δεν μπορούμε να παίζουμε με έναν τομέα που σε αυτή τη θητεία δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την συστημική κρίση που ξέσπασε πριν από λίγο χρόνο και που κυκλικά μπορεί να την ξαναζήσουμε και να τρέχουμε να φτιάξουμε μια νομοθεσία, να διορθώσουμε μια νομοθεσία που δεν θα είναι πλήρης. Σας ευχαριστώ. Δεν... τώρα βλέπω ένα συνάδελφο που θέλει να πάρει το λόγο. Είναι ένα γκίλ. Thank you, Chair. I want Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Περιμένουμε για να ολοκληρώσουμε και την δική μου την έκθεση. Λοιπόν, εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτοί οι θεσμοί είναι κοινωνικού σκοπού. Δεν είναι μόνο δηλαδή χρηματοπιστωτική υπηρεσία. Τα συνταξιωτικά ταμεία, επαναλαμβάνω, έχουν κοινωνικό σκοπό γιατί προέχουν ναι, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αλλά όχι αποκλειστικά. Επίσης είναι σημαντικό όταν κανείς βλέπει την διακυβέρνηση αυτών των οργανισμών να μην το γεμίζουμε μόνο με οικονομολόγους είναι σωστό να πληρούν ε, συλλογικές ε, ε, απαιτήσει, αλλά όχι αποκλειστικά οικονομικοί λόγοι να είναι, γιατί θα πρέπει να σκέφτεται ότι πρόκειται για τη ζωή των ανθρώπων, ότι πρόκειται για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και δεν πρόκειται για καθαρά μαθηματικές εξισώσεις που πρέπει να βγαίνουν. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτά. Ευχαριστώ. Ναι, πολύ Ο ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητέ από την ομάδα μου για την έκθεση αυτή που είναι πολύ καλή για τους λόγους που μόλις εξήγησε και η Νίνα Γκίλ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η συμμετοχή στα ε, προγράμματα των συνταξιδοτικών παροχών είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία και η οδηγία θα πρέπει να μιλάει για το συμπληρωματικό ρόλο των προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά τα προγράμματα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείονται από την κοινωνική ασφάλιση, Δεύτερον, θα δημιουργηθεί, λέμε, ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δήματα ταξιδιωτικών παροχών. Σωστά. Και γι' αυτό και διάφορες τροπολογίες που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα και με την μεταφορά. Ελπίζω να έχουν ληφθεί υπόψη. Έπειτα η συμμετοχή σε τέτοια συνταξιδοτικά ε, προγράμματα δεν πρέπει να παραβιάζει την αρχή ε, της μη διάκρισης εξαιτίας διαφορετικού τόπου κατοικίας, δεδομένου ότι υπάρχει ελεύθερη διακίνηση. Άρα, δεν πρέπει να απαγορεύουμε να χρησιμοποιούνται λογαριασμοί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και να πληρώνονται εκεί οι συντάξεις. Τέλος, κάτι που έχει να κάνει με την ορολογία. ο όρος κράτος προέλευσης ή κράτος υποδοχής δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται αρκετά καλά στην ενιαία αγορά. Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε άλλη ορολογία, την οποία και προτείνω με κάποια μου τροπολογία. Τέλος, η οδηγία αυτή πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να αποφεληθούμε από αυτήν για να πετύχουμε την ε, ενιαία αγορά, να την ολοκληρώσουμε και Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέρφους για τις προσπάθειές τους προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν βλέπω άλλο συνάδελφο να έχει ζητήσει το λόγο, οπότε ο εισηγητής και πάλι για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέρφους που πήραν το λόγο σήμερα εδώ. Αναφέρθηκαν διάφορα ζητήματα και θέλω να απαντήσω τις παρατηρήσεις του Πολ Τάνκ πρώτα απ' όλα, αλλά και σε αυτά που είπε η Νίνα Γκίλ και άλλοι. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για κοινωνικά μέσα, ευρωπαϊκά, για τα οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Συμμετέχουν λίγες χώρες, θα τα καλό να συμμετείχαν περισσότερες. Είναι θετικό ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι πληρώνουν αυτά τα προγράμματα. Και γι' αυτό που είπε η Νίνα, συμφωνώ. Γι' αυτό και κάνουμε αλλαγέ στο κείμενο, ώστε κάθε δικαιούχος να μην έχει ξεχωριστή μεταχείριση. Να είναι κάτι συνολικό. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε την καλή δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα από τους τραστείς. Και σωστά το είπε ο Πολ Τάγκ. Είπε επίσης ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και συμφωνώ. Πολλές φορές ε, απαντάμε μεμονωμένα αναχώρα μέλη στα επίπεδα συνταξιοδότησης. Έτσι κι δεν είναι μια προσέγγιση που κάνει για όλους και θα φαίνεται αυτό στο κείμενο. Σωστά επίσης είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά το ρυθμιστικό αντιτράσμα. Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι ότι θέλουμε ένα βαθμό εναρμόνισης ώστε να μην έχουμε το αρμπιτράζ αυτό. Αν το έχουμε, την επιλογή δηλαδή ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας, είναι γιατί κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετικά το θέμα για το χρόνο, τα ποσά κτλ. Και ακριβώς αυτό είναι που δημιουργεί τη δυσκολία. Να συνεργαστώ με τον Πολ και με άλλους. Κάτι άλλο που ανέφερε είναι ότι πρέπει να υπάρχουν πιο υπεύθυνοι κανόνες, κανόνες για υπεύθυνε επενδύσεις δηλαδή και πιο μακροχρόνιες. Δεν το κι άλλοι. Για τον Ashley Fox αναφέρθηκε στην αναλογικότητα και την επικουρικότητα. Σε οτιδήποτε κάνουμε εδώ δεν μπορεί να επιβάλλουμε επιπλέον κόστος στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα. Δεν πρέπει. Πέρασαν από τη χειρότερη κρίση όλων των εποχών. Χρειάζονται μεγένθηση για να συνεχίσουν. Οπότε το τελευταίο που θέλουμε να κάνουμε είναι να τους επιβάλλουμε επιπλέον κόστος. Ο κύριο Στάγκ έφερε και τι ε, απόψει του για το. Ο κύριο Άσλε συγγνώμη, για το 35 και το αποθετήριο. Υπάρχει θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη γνωρίζω. Για το άστρο 5 θέλω να πω ότι δεν πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ότι η οδηγία δηλαδή θα εφαρμόσεται και σε περιπτώσεις κάτω των 100. Και ευχαρίστω να το βάλω αυτό ξεκάθαρα. Για το 50, για την πλήρη χρηματοδότηση, την απέτηση δηλαδή πλήρους χρηματοδότησης, ναι, όπου υπάρχουν ε, νέα προγράμματα. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ο Άσλι το έχει πει και στις συναντήσεις μας για τις δοκιμές αναλογικότητας μετά τους τριμερείς διαλόγους. Εγώ είμαι ανοιχτό θα χρειαστούμε χρόνο να το συζητήσουμε στις συναντήσεις με τους σκιώδες εισηγητές. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Δεν ξέρω πώς να το λύσω. Οτιδήποτε πάντως βελτιώνει το κείμενο και την εφαρμογή του σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σεβόμενο την αναλογικότητα, είναι ευπρόσδεκτο. Είμαι ανοιχτό. Για τη σημασία της κινητικότητας των Ευρωπαίων εργαζομένων. Σωστά. Γι' αυτό και πρέπει να εξυγχρονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα συνταξιδοτικά ταμεία λειτουργούν, ώστε ένα μεγάλο ποσοστό εργαζόμενων που μετακινείται να καλύπτεται. Αναφερθήκατε επίσης τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Θα το συζητήσουμε και αυτό και θα δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το κείμενο από αυτό. Και σε αυτό είμαι ανοιχτό. Τώρα για τη φαρικιότητα 2, το Solvency 2. Στις τροπολογίες που προτάθηκαν δεν υπάρχει συμφωνία ούτε μεγάλη πλειοψηφία συναδέρφων που να συμφωνεί ότι η Solvency 2 πρέπει να εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση. Και πρέπει να ξέρουμε ότι αν κάποιος προτείνει την επέκταση της όλβανση 2, αυτό σημαίνει επιπλέον κόστος στους ήδη δικαιούχου και μέλη. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Και αν θέλουμε να το στηρίξουμε, να το έχουμε υπόψη μας. Δεν αντικατοπτρίζεται πάντως στις τροπολογίε που έχω πάρει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον Φιλιπ Λαμπέρ για τι παρατηρήσει του έκανε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις από τον Μακάρνη που είναι Καναδός με Ιρλανδικό διαβατήριο όμως. Για αφορολογικούς λόγους έχει το Ιρλανδικό διαβατήριο. Όχι, όχι. Φαντάζομαι ότι αν τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα ήθελε να το έχει. Τέλος πάντων δεν θέλω να απαντήσω. Έχει πάντως Ιρλανδικό διαβατήριο. Και το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για την αρχή της πλήρους χρηματοδότησης. Το στοιχείο κλειδί είναι ο χρόνος που χρειάζεται η κάθε χώρα. Και δεν είναι που παρεμβαίνει το αρμπιτράζ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ισορροπία και όπως είπα και στην αρχή, ευχαρίστως να το κάνω. Συμφωνώ για τη διαφάνεια με αυτά που είπε ο Λομπέρ. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει πού επενδύονται τα χρήματά του που βρίσκονται επενδύσει του. Να ξέρει ποια είναι και η αξιολόγηση κινδύνου. Πώς να πετύχουμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην καλή ποιότητα ρυθμιστικών συστημάτων των χωρών μελών που βρίσκονται πιο μπροστά από εμά. Ευχαριστώ και τον Μαρκοβάλη για τις παρατηρήσεις του. Σωστά είπε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα χρήματα των φορολογούμενων, των επενδυτών και γι' αυτό και χρειάζεται καλύτερη διακυβέρνηση. Και εδώ το στοιχείο κλειδί τελικά στο συμβασμό που θα κληθούμε να κάνουμε πρέπει να δούμε πόσο μακριά θα επεκταθεί η εφαρμογή των ρυθμίσεων των διασυνοριακών IRPs στα εθνικά αντίστοιχα ιδρύματα. Και σωστά επίσης είπε ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας τους κινδύνους που μας περιμένουν Γι' αυτό και έχουν μετροπολογίε του για θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Για την Ινα ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Νομίζω ότι απάντησα και τους στραστής. Έχετε δίκιο. Έχουμε πολύ καλά παλιά προγράμματα με λίγα μέλη και δικαιούχους. Πρέπει να είμαστε σίγουροι με τις δοκιμές αναλογικότητας που κάνουμε ότι δεν θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο που δεν τους μεταχειρίζεται σωστά. Ευχαριστώ και τον κύριο Φερνάντες για τις δικές του παρατηρήσεις. Όντως έχει υποβάλει ενδιαφέρουσες τροπολογίες που θα τις μελετήσουμε στις συζητήσεις που θα έχουμε με τους σκιώδες. Ωραία, νομίζω ότι απάντησα στις παρατηρήσεις των συναδέρφων και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να μας καλύπτει όλους μέσω των τροπολογιών που υποβλήθηκαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Μπράιαν. Χρονοδιάγραμμα. Μετά από επιτυχείς διαπραγματεύσεις, η ψηφοφορία θα γίνει την πρώτη 12 για την Ολομέλεια προβλέπεται να φτάσει τον Ιανουάριο του 2016. Έχετε λοιπόν ε, υπόψη όλοι και όλες ότι 1η Δεκεμβρίου προβλέπονται πολλές ψηφοφορίες. Ελπίζω ότι θα προλάβουμε. Περιμένοντας τώρα τους κυρίους Ντάισελμπλουμ και Ρέγκλινγκ θα κάνω μια σύντομη διακοπή μέχρι ότου φτάσουν.

Ναι, το Ζάγκε τελειώνει. So hello everybody. Please take a seat. Ο πρόεδρος Φέρμπερ, σας παρακαλώ καθίστε. Κάποια στιγμή ανησυχήσαμε μήπως ε, χάθηκαν οι ομιλητές μας, αλλά βρεθήκαμε. Οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ελπίζω ότι δεν ε, διετάραξαν το πρόγραμμά σας. Σας περιμέναμε. Καλώς ε, ήρθατε, με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Ευρωομάδας, κύριο Ντάισελμπλουμ και τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας κ. Ρέγκλινγκ για ανταλλαγή απόψεων για το νέο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάδος. Προβλέπετε να ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα προγράμματα προσαρμογής σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Εμείς λοιπόν η Επιτροπή Οικονομικών είμαστε η αρμόδια επιτροπή για την διεξαγωγή του διαλόγου. Το τρίτο οικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδος άρχισε με υπογραφή του ε, Μνημονίου Συμφωνίας στις 18 Αυγούστου και συνεχίζεται μέχρι 18 Αυγούστου του 2018. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει 25 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και κόστη για την ενδεχόμενη ε, διάλυση τραπεζών. Ε, προβλέπεται και ένα ποσό από τον EFSM που περιλαμβάνεται στο ίδιο συνολικό ποσό. Το μνημόνιο προβλέπει τέσσερις πυλώνες. Αποκατάσταση της βιωσιμότητας του φορολογικού συστήματος, αύξηση της ανταγωνιστικότητας ε, ε, της οικονομίας και ε, αναδιάθρωση του κρατικού μηχανισμού. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε Πρόεδρε της Ευρωομάδας και εσείς και διευθυντά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ε, θα προβείτε σε σύντομες δηλώσεις και μετά θα προχωρήσουμε σε ανταλλαγή ερωτήσεων-απαντήσεων. Αρχίζουμε με τον κύριο Ντάισελμπλουμ, πρόεδρο της Ευρωομάδας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Καλησπέρα. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και ζητώ συγγνώμη που χρειάστηκε να ακυρώσω έναν προηγούμενο διάλογο που είχαμε προβλέψει για την 22η Σεπτεμβρίου. Αυτό έγινε εξαιτία των θεμάτων για τη μετανάστευση με τα οποία έπρεπε να ασχοληθώ τότε και γι' αυτό ακύρωσα τη συνάντησή μας εκείνη. Σήμερα το απόγευμα ήμασταν ε, δίπλα. Περιμέναμε να έρθει κάποιο να μα πάρει για να έρθουμε εδώ. Γι' αυτό δεν ήρθαμε γρήγορα στην αίθουσα. Ήμασταν όμω εδώ δίπλα. Περιμέναμε να έρθει κάποιο να μα πάρει και να μα συνοδεύσει εδώ. Και εμεί ανησυχούσαμε γιατί είχαμε ξεμείνει. Λοιπόν, έρχομαι στο θέμα τη Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να αναφέρω διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, κοιτώντα τι έχει γίνει μέχρι τώρα, πού βρισκόμαστε σήμερα και κυρίω προ τα που πάμε. Η προηγούμενη χρονιά ήταν ε, γεμάτη προκλήσεις πάνω απ' όλα για τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι πέρα από τα οικονομικά και κοινωνικά τους προβλήματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν και μια μεγάλη περίοδο αβεβαιότητας. Τεράστιες προσπάθειες και θυσίες που έκαναν τα τελευταία χρόνια για να επιστρέψει η χώρα του σε βιώσιμη ανάπτυξη κινδύνευσαν να πάνε στράφη. Η διαδικασία διαπραγματεύσεων ήταν μακρά και δύσκολη. Μερικές φορές μάλιστα περίχε και διάφορες εκπλήξεις. Υπήρχαν και πιο εύκολοι τρόποι για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει τελικά καταλήξαμε σε συμφωνία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καταλήξαμε λοιπόν σε ένα νέο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Ο δικός μου στόχος και των άλλων υπουργών στο Eurogroup ήταν να διασφαλίσουμε ένα μέλλον γεμάτο ευημερία για την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τη δέσμευση τη δικιά μου και των υπολείπων επ' αυτού. Θέλουμε να συνοδεύσουμε την Ελλάδα στις προσπάθειες που κάνει για μεταρρύθμιση προκειμένου η οικονομία της να μπει και πάλι στον δρόμο της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Πριν από ένα χρόνο όμως, με την πέμπτη και τελευταία ε, αξιολόγηση του δεύτερου μνημονίου, οι προοπτικές τη Ελλάδας φαινόντουσαν αρκετά καλές. Η οικονομία προχωρούσε προς την ανάπτυξη και το δεύτερο εξάμεινο του 2014 μετά από μεγάλη ύφεση και τα κρατικά ομόλογα πήγαιναν καλύτερα. Όμως παρά το γεγονός ότι αποφάσισε για δύο μήνες παράταση του προγράμματος αυτού το Eurogroup τελικά δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση έγκαιρα και χρειάστηκε επιπλέον παράταση. Έπρεπε να γίνει πολλή δουλειά μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα για να επανέλθουμε σε βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Ξέπνευσε τελικά το πρόγραμμα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε ότι δεν μπορεί να αυξήσει το όριο του ELA και χρειάστηκαν ε, capital controls. Είμαι πεπισμένος και το έχουμε πει ξανά και ξανά ότι θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι. Πάντως σε αυτά τα πλαίσια, τελικά στις 12 Ιουλίου, μετά από έντονη δουλειά στο Eurogroup, άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για ένα νέο φιλόδοξο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, μια από ένα τέτοιο πρόγραμμα στο μεταξύ ζήτησαν οι ελληνικές αρχές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πιστεύω ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα προσαρμογής είναι καλό για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη. Μετά από ένα διέξοδο πολλών μηνών, φάνηκε η πολιτική βούληση όλων των πλευρών να διατηρηθεί η ακαιρεότητα της ε, Ευρωζώνης. Και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Η Ελλάδα και το μέλλον της βρίσκεται μέσα στην Ευρωζώνη. Με τις προηγούμενες δράσεις το πρόγραμμα έχει ένα σκέλος ε, προκαταβολών και είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί πιστοσύνη. Είναι ισορροπημένο το πρόγραμμα. Περιλαμβάνει ήπια μέτρα προσαρμογή. Χρησιμοποιούνται καλύτερα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη βραχοπρόθεσμα. Κάτι το οποίο οδηγεί βέβαια στην ανάγκη για φιλόδοξες ε, μεταρρυθμίσεις επιγόντως. Το πρόγραμμα επίσης βασίζεται στα επιτεύγματα των προηγούμενων ετών. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βάζουν τα συμφέροντα των καταναλωτών και των εργαζόμενων πριν από τα παγιωμένα συμφέροντα. Και θέλουμε έτσι να βοηθήσουμε να εξυγχρονιστεί το ελληνικό κράτος και η οικονομία να είναι πιο ανταγωνιστική και πιο παραγωγική στα διεθνή πλαίσια. ίδια πλαίσια θέλω να τονίσω ότι είναι ζωτική σημασία. Ζωτική σημασία, επαναλαμβάνω, η νέα ελληνική κυβέρνηση να ενστερνιστεί τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις και να προχωρήσει σε αυτό το τομέα προκειμένου να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη λειτουργία του κράτους και στην ικανότητα της οικονομίας να δημιουργήσει ευημερία για όλους. Πρέπει να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, η διαφθορά, να υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύστημα φορολόγησης. Όλα αυτά πρέπει να παγιωθούν. Η τεχνική αρρωγή υπάρχει για να στηριχθεί ακριβώς αυτή η διαδικασία. Με δύο λόγια, το πρόγραμμα αυτό θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα προκειμένου η Ελλάδα να επιστρέψει σε έναν δρόμο ισορροπημένη και δίκαια ανάπτυξη αλλά και σε δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Τώρα, στρεφόμενο προ το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 31 Οκτωβρίου δημοσίευσε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ελληνικού τραπεζικού τομέα και εντόπισε ένα κενό 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι τράπεζε την προηγούμενη εβδομάδα υπέβαλαν τα σχέδιά του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το πώ θα καλύψουν το κενό αυτό μέχρι τα τέλη τη χρονιά. Το μέγεθο του κενού αυτού τελικά είναι λιγότερο από ό,τι αρχικά είχαν ε, προβλέψει κάποιοι τουλάχιστον από εμάς πριν από μερικού μήνε. Και αυτά δεν είναι καλά νέα για τις τράπεζες, αλλά και για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Και έτσι οι τράπεζες θα μπορέσουν να καλύψουν, αν όχι όλο, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του κενού αυτού μέσω ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να δανειστούν επιπλέον ε, κονδύλια για την ανακεφαλοποίηση των ε, τραπεζών πέρα από τα 10 δισεκατομμύρια τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα. Σήμερα οι αρχές εφαρμόζουν τα προαπαιτούμενα. Χτες στο Eurocrop σημειώσαμε τις τελευταίες εξελίξεις και καταλήξαμε στο τι πρέπει να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών μέσα σε επόμενες εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πρόοδο προκειμένου να υπάρξει ένα πλαίσιο για, την, ε, για τη, τα δάνεια για τις κατοικίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να διώξουμε τους ανθρώπους από τα σπίτια τους, αλλά πρέπει να μειωθεί το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να εξηγιανθεί και πάλι ο ελληνικός τραπεζικός τομέας. Υπάρχουν λοιπόν τα προαπαιτούμενα για τις τράπεζες. Και είναι ζωτική σημασία. Οι ελληνικές αρχές θα καλύψουν τα προαπαιτούμενα μέσα, σε μέσα στην εβδομάδα αυτή. Και μόνο τότε θα μπορέσει η υποδόση να εκταμιευθεί και να μεταφορθούν τα χρήματα που χρειάζονται για την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών